εξέλιξη η συζήτηση, αύριο θα γίνει ψηφοφορία. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, στην κοινή συζήτηση για τα σήματα, για τα εμπορικά σήματα. Η Κεκυλία Βίξτρομ και μετά για τις νομοθεσίες των κρατών μελών περί σημάτων. Επίσης Κεκυλία Βίξτρομ. Η εισηγήτρια πρώτα επί τέσσερα ολόκληρα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είχα την τιμή να είμαι εισηγήτρια στο πακέτο για τα εμπορικά σήματα από την Άνοιξη του 2012 και με αυτή την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τους βοηθούς στο Κοινοβούλιο και στο, στην Κομισιόν και να ευχαριστήσω θερμά και τις ε, πολυάριθμες προεδρίες που εργάστηκαν κυρίως η Ιταλική και η Λετωνική Πρόεδρια που έκαναν εξαιρετική δουλειά στις πιο κρίσιμες φάσεις των διαπραγματεύσεων. Τώρα θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στα επιτεύγματα αυτού του φακέλου. Οι μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στους, τριμερί, στους διαλόγους ε, σημαίνουν ότι οι εταιρείε έχουν ταχύτερη πρόσβαση σε εμπορικά σήματα και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς συμβιβασμού στην ποιότητα των Τι Ξυγχρονίστηκαν οι διοικητικές διαδικασίες σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και θα δούμε αυξημένη εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων ε, στα πλαίσια των ε, βελτίστων πρακτικών. Τώρα, το, η νομοθεσία αυτή καθ' αυτή, ε, έχουμε εξυγχρονίσει πολλές διατάξεις που λαμβάνουν υπόψη τεχνολογικές εξελίξεις και προσθέσαμε και σημαντικές διασφαλίσεις ε, ό,τι αφορά τη χρήση παράτυπα των εμπορικών σημάτων για διάφορους λόγους, ε, για καλλιτεχνική έκφραση ή ε, παραχάραξη. Θέλω να ευχαριστήσω ένα παλιό συνάδελφο από τη Σουηδία, που επέστησε την προσοχή μας όλα αυτά. Παλιός συνάδελφος δεν είναι πια μαζί μας. Μπορεί να έχετε κάποιοι από εσά λάβει επιστολές από μη κυβερνητικέ οργανώσεις την προηγούμενη εβδομάδα που εκφράζουν ανησυχίες σε ό,τι αφορά τα γενώσιμα και την μεταφορά τους σε αναπτυσσόμενες χώρες. Θέλω να υπογραμμίσω την θέση μας και ε, τα γεγονότα. Μπορώ να διαβεβαιώσω όλους ότι επουδενή δεν θα υπάρξει πρόβλημα για το, ε, την ε, διαμετακόμιση ε, γενοσύμων σε αναπτυσσόμενες χώρες λόγω αυτής της νομοθεσίας. Όλη μου τη ζωή έδινα μάχη για την ανάπτυξη και ποτέ μα ποτέ δεν θα επέτρεπα ένας νόμος με το όνομά μου να εμποδίζει τους ανθρώπους στις αναπτυσσόμενες χώρες από την πρόσβαση στα φάρμακα. Αυτό είναι βέβαιο. Η φιλοδοξία μας ήταν κοινή σε όλη την κοινοβουλευτική διαπραγματευτική ομάδα. Είμαστε ενωμένοι πάνω σε αυτά και ε, επίσης, όπως σας είπα, ε, βάλαμε κάποιες ρήτρες ε, διασφάλισης πολύ ισχυρές. Και εδώ, εις ό,τι αφορά τη διαμετακόμιση των γενοσύμων αυτά αφορούν ε, όχι τα εμπορικά σήματα αλλά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Είμαι περήφανη σήμερα διότι επιτύχαμε ισορροπία μεταξύ καταπολέμησης οργανωμένου εγκλήματος και τη, τα, καταπολέμηση των ε, παραχαραγμένων προϊόντων. Υπογραμμίζω ότι δεν υπάρχει κίνδυνο σύγχυσης μεταξύ γενώσιμων και παραχαραγμένων ε, φαρμάκων, ε, ε, λάθος φαρμάκων. Όλες οι χώρες καταπολεμούν τα τελευταία και βεβαίως εις ό,τι αφορά την νομοθεσία για τα για τους δασμούς προβλέπονται και ποινικέ ρήτρε σε περίπτωση παράβασης. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες σε μια σημαντική μάχη πολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος που πλήττει τους πιο ευάλωτους. Εδώ είμαστε ενωμένοι όλοι. Θα επανέλθω και αργότερα, αλλά περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Πρόεδρε, τη συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπιενκόφσκα, η Επίτροπος, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, πρώτα-πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμό την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και επίσης να συγχαρώ την εισηγήτρια την κυρία Δίξτρομ για ε, αυτήν την ε, έκθεση για το πακέτο αυτό το νομοθετικό πρόκειται για πάρα πολύ ε, επικοδομητικό ε, πνεύμα το οποίο επεκράτησε μετά από δύο χρόνια καταλήξαμε σε μια συμφωνία ήταν περίπου και συζητήσεις είναι τεχνικό το ζήτημα και αυτού του είδους ε, η μεταρρύθμιση για το εμπορικό σήμα είναι σημαντικό για την καινοτομία ε, και για την ανταγωνιστικότητα. Οπότε τώρα θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και την ανάπτυξη και την καινοτομία και θα υπάρχει ένα σύστημα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση προσβασιμό ε, για όλες τις επιχειρήσεις. Θα έχουμε πιο συγκρατημένες δαπάνες, ταχύτητα, προβλεψιμότητα και θα υπάρξει και ασφάλεια δικαίου. Οπότε το, το, τα κέρδη είναι ξεκάθαρα για όλους, γιατί έτσι θα έχουμε σημαντικά προς και περαιτέρω εναρμόνιση του δικαίου σημάτων στην Ένωση. Τώρα να σας τονίσω ε, κάποια σημεία από τα ωφέλη που θα έχουμε πρώτα-πρώτα. Αυτές οι μειώσεις που συμφωνήθηκαν θα οδηγήσουν μέχρι 40% εξοικονόμηση δαπανών, ιδίω για τι επιχειρήσει οι οποίε θέλουν να υπάρξει ε, προστασία πέραν τη αρχική δεκαετία. Δεύτερον, η μεταρρύθμιση τη οδηγία θα μα οδηγήσει σε περισσότερη ένταξη τη πολιτική ε, πέραν των παλαιών υπηρεσιών προστασία σημάτων. Επίσης θα υπάρξουν ε, λιγότερο επαχθείς διαδικασίες και γραφειοκρατικές, θα ωφελήσουν κυρίως τις ΜΜΕ και θα υπάρξει ε, προστασία καλύτερη για τα σήματα. Επίσης θα έχουμε στο μέλλον διαδικασίες διαβούλευσης αλλά και προσφυγής. Αυτά είναι δείγματα της βελτίωσης που θα υπάρχει επίσης η ε, δικαιούχοι σημάτων θα μπορέσουν κλίτρα να καταπολεμήσουν τις ε, απομιμήσεις ε, ιδίω τις περιπτώσεις που αυτά τα παράνομα προϊόντα διαμετακομίζονται στη μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ε, θα γίνουμε επομένω ένας ε, κόμβος για την ε, διανομή και την εμπορία αυτών των προϊόντων. Οπότε όλα αυτά θα οδηγήσουν σε ενθάρρυνση του νομίμου εμπορίου και επίσης θα έχουν περισσότερη ασφάλεια δικαίου όταν μπορέσουμε να προσαρμόσουμε αυτό το δίκαιο σημάδων στο μοντέρνο εμπόριο και επίση όταν ξεκαθαριστούν τα όρια της προστασίας των σημάτων σε σχέση τώρα με, τη, με τον κανονισμό και όσον αφορά τον ορισμό ε, του διευθυντού ε, της υπηρεσίας του Αλικάντε ο οποίος θα ε, διεκπεριώνει τα, του δικαίου των σημάτων που θα δεσπιστεί τώρα θα σας πω ότι εδώ υπάρχει κάποια συμβατότητα σε σχέση με τα όσα προβλέπονται ε, από τον κανονισμό για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Βέβαια παρόλα αυτά έχουμε κάποια σημαντικά σημεία των προτάσεων Κομισιόν ε, τα οποία δεν τα <clears throat> εγκρίνεται οπότε το τελικό κείμενο του κανονισμού παρόλα αυτά πρόκειται να επιφέρει καλύτερες βελτιώσεις όσον αφορά τη λογοδοσία ε, αυτής της υπηρεσίας. Οπότε αυτό θα ολοκληρώσει τον συμβασμό που κλείσαμε και που τον χαιρετήσουμε και έτσι θα ολοκληρωθεί αυτή η δέσμη νομοθετικών μέτρων. Σας ευχαριστούμε και εμείς ε, κυρία Επίτροπε, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα δώσουμε το λόγο στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Πρώτα-πρώτα ο κύριος Πάβελ Σβόποντα για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Νομικής Επιτροπής που έλαβαν μέρος σε αυτή την μεταρρύθμιση και επίσης ε, την εισηγήτρια. Και η προστασία των εμπορικών σημάτων είναι ένα πολύ σημαντικό έργο και συμφωνήσαμε ε, ως προς τις αλλαγές ε, της υπάρχουσας της ισχύας νομοθεσίας που θα έχουν θετικές επιπτώσεις για όσους ασχολούνται με την προστασία των εμπορικών σημάτων. Ε, αυτό, και αυτό δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις. Γνωρίζω ότι οι τροπολογίες που προτάθηκαν προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία και να είναι λιγότερο δαπανηρή, ε, θα διευκολύνει επίσης τους χρήστες. Επίσης, και οι άλλες αλλαγές που πηγάζουν από της τη Λισαβόνα αποδεικνύει ότι μπορούν να γίνουν πρακτικές αλλαγέ, οι οποίες όμως δεν είναι πάντοτε κατανοητές στο ευρύ κοινό. Συμφωνώ με τις προτινόμενε αλλαγέ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, εξ ονόματος των σοσιαλιστών, ε, σας δίνω 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Το πακέτο για τα εμπορικά σήματα είναι πάρα πολύ σημαντικό στην καταπολέμηση των πλαστών προϊόντων. Διαπιστώνουμε πως ε, έχει μεγάλη σημασία ε, το θέμα αυτό. Ήδη λειτουργεί ένα σύστημα ευρωπαϊκών εμπορικών σημάτων αρκετά καλά. Με το νέο σύστημα όμως έχουμε αρκετές ε, βελτιώσεις και ελπίζουμε να οδηγηθούμε σε μεγαλύτερη καινοτομία και ανάπτυξη. Τι έχουμε λοιπόν, έχουμε νέα μείωση των ε, τελών, καλύτερη συνεννόηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας και των Εθνικών Γραφείων ε, και η καταχώρηση ενός Ευρωπαϊκού Εμπορικού Σήματος. Ανέφερε επίσης κάτι σημαντικό η κυρία Βίξτρομ, το οποίο είναι και για εμάς σημαντικό. Δηλαδή μπορούμε να εγγυηθούμε πως θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμα τα γενώσιμα στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Κάτι το οποίο βεβαίως πρέπει να μας απασχολεί να είναι διαθέσιμα τα γενώσιμα σε όλες τις ε, χώρες ε, και βεβαίως θα υπάρχει και το θέμα της ε, ελεύθερης έκφρασης τη γνώμης, το οποίο μόνο ως παροδία μπορώ να θεωρήσω ότι εμποδίζεται από ένα τέτοιο κανονισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ΚΟΕ. Ο κύριος Μαστάλκα για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητή Σεσίλια. Ο στόχος ε, των ευρωπαϊκών εμπορικών σημάτων είναι να διακρίνουμε μεταξύ των προϊόντων στην αγορά και να μπορούν έτσι οι καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα και υπηρεσίες ε, αυτά τα οποία ακριβώς θέλουν όμως. Το σύστημα αυτό θα λειτουργήσει παράλληλα με τα εθνικά συστήματα προστασίας. Ε, δεν θα είναι ανταγωνιστικό αλλά συμπληρωματικό. Οπότε έχουμε νομίζω ένα καλύτερο μέσο καταπολέμησης των πειρατικών ε, πλαστών προϊόντων. Και οπωσδήποτε με μια ενιαία καταγραφή δίνεται πλέον ένα εμπορικό σήμα το οποίο θα έχει ίση προστασία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονό πως έχουμε πανευρωπαϊκή νομοθεσία αντί για 28 εθνικούς νόμους δίνει μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα και βεβαίως μειώνεται και το κόστος της νομοθεσίας και των νομικών υπηρεσιών. Άρα η διαδικασία αυτή γίνεται φτηνότερη. Επίσης σημαντικό το ότι βρήκαμε θετικές λύσεις με όλους τους άλλους σκιώδεις εισηγητές και σας ευχαριστώ και σας αγαπητοί και κοιλία για τα φάρμακα και καλά Χριστούγεννα σε όλους. Σας ευχαριστώ για τους πράσινους. Ο κύριος Μαξ Άντερσον για 2,5 λεπτά έχετε το λόγο. Eh, ευχαριστώ πρώτα πρώτα την εισηγήτρια την κυρία Βίξτρομ αλλά να ευχαριστήσω και τους κοιόδης εισηγητές. Επρόκειτο για το πρώτο θέμα το οποίο με επισχόλησαν στα πλαίσια του τριμμένου διαλόγου. Και πρέπει να σα πω ότι εντυπωσιάστηκα από το έργο που επιτελέσει την πρώτη για αξιολογή έκθεση, γιατί αυτό το οποίο θέλουμε τώρα να έχουμε ένα πιο ευελικτό σύστημα και είπαμε ότι θα εξοικονομούμε όλες αυτές τις ε, δαπάνες που ε, απαιτούνται μέχρι σήμερα. Επομένω υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία σε αυτό το νομοθέτημα. Όμω, όσον αφορά την ελευθερία έκφραση, για εμά του πράσινου, εμάς, ε, αυτό μας απασχολεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στην έκθεση. Επίσης, ε, μας απασχολεί το θέμα των φαρμάκων, των γενοσύμων. Εμείς ασχοληθήκαμε επί πολύ χρόνο με το θέμα αυτό και είχαμε πολλές επιφυλάξεις για την ε, στάση του Συμβουλίου. Έχουμε επίσης και από τους γιατρούς χωρί σύνορα μια επιστολή που αφορούσε ακριβώς το τι θα γίνει με αυτά τα φάρμακα για τα οποία δεν παρέχονται αρκετές εγγύσει. Οπότε επίση υπάρχει ο κίνδυνο εδώ αυτά τα γενώσιμα δεν θα καλυφθούν. Θα πρέπει βέβαια να ελέγχει στον παιδί αυτό ο κίνδυνο, αλλά εμεί οι πράσινοι θεωρούμε ότι δεν σημειώθηκε αρκετή πρόοδο. Εμεί δώσαμε αγώνα ούτω ώστε να αποσπάσουμε περισσότερε εγγύσει. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Θα καταψηφίσουμε. Η πρόταση γιατί για εμά το τι θα γίνει τα γυμνασμένα φάρμακα είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Και τώρα για το EFTD. η κυρία Φεράρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ να αρχίσω ευχαριστώντας την εισηγήτρια, την συνάδελφο Βίξτρομ για τις προσπάθειες που κατέβαλε αλλά και τους σχεδόν ηγητές. Είναι πολύ σημαντικό το σύστημα για το παρικό σύστημα της Ευρώπης και επίσης για κάποια άλλα εθνικά ή υποσυστήματα όπως ας πούμε για το Ιταλικό σύστημα. Εκεί που το made το οποίο είναι συνώνυμο της ένδειξης ε, προέλευσης είναι εγγύηση κατά των παραπίσεων και απομίσεων. Οπότε ε, νομίζουμε ότι χωρίς δυσκολία θα περάσουν αυτές οι διατάξεις για το σήμα στην Ευρώπη. Επίσης να έχουμε και τη σχετική ε, ρήτρα, τη φέργιου σου, ώστε θέλουμε να υπάρχει ερμηνεία των κανόνων ε, για την αποκλειστική χρήση. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε σε σχέση με την καλλιτεχνική δημιουργία. Επίσης, ε, νομίζουμε ότι η σχετιολογική έκδοση σε καλά τα λέω τα θεμελιώδη δικαιώματα και να προσέξουμε τι θα γίνει με την ελευθερία της έκφρασης και επίσης να δούμε τι θα γίνει με την ελεύθερη διαμετακόμιση των ε, γενοσύμων. Δεν θα πρέπει να ε, μην κάνουμε τίποτα, ούτως ώστε να, να, να την πορεία των απομίσεων των φαρμάκων, κάτι που είναι πάρα πολύ πιο για την υγεία των Ευρωπαίων. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Φεράρα, λέει ο πρόεδρο. Και ο κύριος Σβιέφκα για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, όλη αυτή η διαδικασία για τη μεγάλη μεταρρύθμιση χρειάστηκε περίπου τρία χρόνια. Η Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων αλλά και άλλοι ευρωβουλευτές ασχολήθηκαν με αυτό το κείμενο για να γίνουν οι αναγκαίε αλλαγέ προκειμένου να υπάρξει προστασία των εμπορικών σημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τελική επιτυχία βεβαίως ε, οφείλεται πολύ ε, στην εισηγήτριά μας η οποία φρόντισε να υπάρχουν διατάξεις σαφείς και αρχές σαφέστατες για τους χρήστες. Πράγματι πρόκειται για μεγάλη επιτυχία. Εδώ μιλάμε για προϊόντα που προκύπτουν από παραποίηση, αλλά υπάρχουν και άλλες αλλαγές, όπως ε, ευκολότερη καταγραφή και εγγραφή των εμπορικών σημάτων, υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια του Μητρώου των Εμπορικών Σημάτων, Επίσης πώς γίνεται η άρνηση μιας εγγραφής. Ε, το σημαντικότερο όμως είναι ότι αυτές οι νέες αρχές θα είναι αποτελεσματικές στην πράξη. Διότι αν δεν είναι αποτελεσματικές οι νέες αρχές, τότε η επιτυχία δεν θα είναι πλήρης. Οι διατάξεις αυτές θα μας επιτρέψουν καλύτερη συνεργασία, για παράδειγμα μεταξύ ε, των αρμοδίων οργάνων ε, για τα ε, διπλώματα βρεσιτεχνίας στα διάφορα κράτη-μέλη. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για την επιτυχή εφαρμογή αυτού του εγγράφου που έχει ως αντικείμενο πιο συγχρονισμένο σύστημα των ευρωπαϊκών σημάτων. Η Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων αντιμετώπισε με ευρύτητα αυτό το θέμα και ολοκληρώνεται όλη η εργασία που γίνεται. Επίσης πρέπει να γίνει μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων τεχνίας και πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και από τυπική άποψη όμως θα ήθελα να σας πω ότι είναι απαράδεκτο τη στιγμή όπου γνωρίζουμε εδώ και καιρό ότι στις 7 η Νομική Επιτροπή έπρεπε να συνεδριάσει για να γίνει ανταλλαγή απόψεων το, ο, σχεδιασμ, ο προγραμματισμός της Ολομέλειας δεν το έλαβε υπόψη και ε, εκ παραλίλου με αυτή τη συζήτηση γίνεται και η συζήτηση στην Ολομέλεια. Γι' αυτό παρακαλώ να φροντίσετε να μην υπάρχουν τέτοιες επικαλύψεις στο μέλλον. E, Παρακαλούμε να μην ξεπεράσετε το χρόνο μιλίας σας στο μέλλον. Θα διαβιβάσω το έτοιμά σας στους συναδέλφους. Μια πληροφορία για όλους τους συναδέλφους από την Ουγγαρία και την Πολωνία. Πριν από λίγο ε, έχουμε τα αποτελέσματα του αγώνα. Η Πολωνία νίκησε. Μιλάμε για το μπάσκετ γυναικών. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Νεγκρέσκου. Ο εξυγχρονισμός του συστήματος ε, εμπορικών συμμάτων θα πρέπει να οδηγήσει σε λειτουργία του συστήματος ε, και στην καταπολέμηση της ε, πειρατείας που κοστίζει τεράστια ποσά και βλάπτει και τους καταναλωτές. Βεβαίως ο στόχος μας εδώ πέρα έχει σχέση και με την υγεία αλλά και με τα θεμελιώδη δικαιώματα και χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να μειώσει τη γραφειοκρατία, να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και να μειώσει το κόστος κατά 37%. Με τους ε, νέους ε, κανονισμούς μειώνονται οι εξαιρέσεις ε, και βεβαίως ρυθμίζονται καλύτερα τα προϊόντα τα οποία είναι καθοδόν. Και βεβαίως ε, θα πρέπει να δούμε το τι γίνεται με τους αρμόδιους φορείς και τα έσοδά τους, καθώς θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων για να αποδίδει και το σύστημα. Δυστυχώς στη Ρουμανία συχνά υπάρχει παραπλάνηση των καταναλωτών με πλαστά και πειρατικά προϊόντα και πρέπει λοιπόν να γίνουν εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών και των εταιριών, ε, κυρίως των μικρομεσαίων, που θέλουν να διασφαλίσουν τα εμπορικά τους ε, σήματα. Ένα κοινό σύστημα βεβαίως ε, θα βοηθήσει την ευρωπαϊκή οικονομία σε σχέση με τους ανταγωνιστές της ε, και θα πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος στην Ευρώπη και στη Ρουμανία ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Νταμπάσκι έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω, έχω, έχω. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επιτυχή κατάληξη της ε, διαπραγμάτευσης. Να ευχαριστήσω την κυρία Βίξτρομ και τους ε, σκιώδεις εισηγητές για την πολύ καλή δουλειά που έκαναν. Έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν μπορούμε παρά να επενέσουμε. Έχουμε όμως και μία ανησυχία γιατί γίνεται μία αναφορά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Μιλάμε για ένα κονδύλιο το οποίο έχει βγει για να καταπολεμηθούν παραβιάσεις ε, των πνευματικών δικαιωμάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να προστατευθούν ακριβώς ε, τα δικαιώματα, αλλά στο εθνικό επίπεδο νομίζω λαμβάνονται καλύτερα αυτές οι αποφάσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Τώρα λοιπόν... Περνάμε στη διαδικασία του KSDI. Ο κύριος Αλπόποβιτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο και ευχαριστώ επειδή τα πολωνικά εμπορικά σήματα θα παραμείνουν πολωνικά. Ευχαριστούμε πολύ για το έγγραφο και την έκθεση, ε, κυρία Βουλσκρόμ. Πράγματι, έχετε να κάνετε με το δύσκολο θέμα της παραποίησης και ε, με την εξασφάλιση της πιστοποίησης και της ανταγωνιστικότητας. Αυτά είναι πολύ δύσκολα θέματα. Αφενός είναι δύσκολο να βρείτε πώς γίνεται η παραποίηση και από την άλλη είναι δύσκολο να απλουστεύεται η νομοθεσία. Πιστεύω ότι μια καλύτερη προσέγγιση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σημαίνει καλύτερη διερεύνηση ε, των αιτίων ε, που εμποδίζουν την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Okay. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το σύστημα προστασίας των εμπορικών σημάτων θα πρέπει να είναι απλό, φθηνό και αρκετά ευέλικτο, έτσι ώστε να παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε προστασία που αντιστοιχεί στις ανάγκες τους. Για παράδειγμα, ορισμένοι χρήστε επιθυμούν προστασία μόνο σε ένα κράτο μέλο, ενώ άλλοι επιθυμούν ενιαία προστασία και στα 28 κράτη-μέλη τη Ένωση γι' αυτό το λόγο πρέπει να διατηρηθεί παράλληλα η προστασία των εμπορικών σημάτων σε εθνικό επίπεδο. αυτό σημαίνει εμπέδωση μιας συμπληρωματικής σχέσης μεταξύ του ενωσιακού και των εθνικών συστημάτων προστασίας εμπορικών σημάτων. στο πλαίσιο αυτό πρέπει να κατοχυρώνεται η αρχή της εδαφικότητας η ασφάλεια του δικαίου και η σαφήνεια τόσο σε περίπτωση ομοιότητας όσο και σε περίπτωση χρήσης ταυτόσιμου σήματος για ταυτόσιμα προϊόντα ιδιαίτερη μέρημνα πρέπει να δοθεί για την διευκόλυνση κατοχύρωσης και προστασίας του εμπορικού σήματος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν χτυπηθεί από την οικονομική κρίση και την λιτότητα ιδίως στην ελλάδα και στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου. ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Ε, gospodine predsjedavajući e, želim vas upozoriti na jedan problem kojega ćemo uskoro imati. θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας επί ενός προβλήματος το οποίο θα εμφανιστεί σύντομα. Δηλαδή, όταν θα υιοθετήσουμε τις αποφάσεις που έχουν σχέση με την ε, γεωργία και θα έχουμε το ευρωπαϊκό μας σήμα το οικολογικό μας σήμα για τα βιολογικά προϊόντα. Θα υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση στη, ανάλογα με τα ευρωπαϊκά προϊόντα, όπου το σήμα δεν θα θεωρείται ότι πρόκειται για βιολογικό προϊόν πανομοιότυπο μεταξύ των χωρών. Δηλαδή, θα αναφέρεται διαφορετικά το εντομοκτόνο, για παράδειγμα, ε, μεταξύ των χωρών και πώς θα γνωρίζουμε ότι πρόκειται για πανομοιότυπο βιολογικό προϊόντο. Αυτό μπορεί ε, να ε, οδηγήσει σε παρερμηνίες ε, και δεν θα γνωρίζουμε ποια είναι η φύση του προϊόντος. Κυρία Επίτροπος, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα προσεκτικά τις ε, παρατηρήσεις σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συνεισφορά σας στην συζήτηση αυτή. Να αναφέρω πρώτα κάποια σημεία κλειδιά. Πρέπει να τονίσουμε πως οι κλάδοι οι οποίοι εξαρτώνται κατά πολύ από τα εμπορικά σώματα συνεισφέρουν πάρα πολύ στην ευρωπαϊκή οικονομία. Και άρα με το να συμφωνήσουμε σε ένα αποτελεσματικότερο νομικό πλαίσιο, οπωσδήποτε θα βοηθήσουμε την ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα. Επίσης θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τα πλαστά προϊόντα για να σταματήσουν επίσης οι συνέπειες που έχουν αυτά στην υγεία, βέβαια και στην καινοτομία και στην ανάπτυξη και σημαντικό είναι να σημειώσουμε πως ε, ο συμβιβασμός αφορά μόνο τα εμπορικά σήματα. Δεν έχει ούτε μία σχέση με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τα γενώσιμα φάρμακα. Παρόλα αυτά, το πακέτο αυτό έχει κάποιες ε, διασφαλίσεις για να υπάρχει μία ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα. Το αναφέρατε μερικοί. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω και να ζητήσω την στήριξή σας για να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα για τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να κάνει οικονομικές ε, μεταρρυθμίσεις. Ενισχύοντας ε, την κοινοτομία και την ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε. Για να ολοκληρωθεί η συζήτηση, δίνω τον λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Βίξτρομ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας αναφέρω κάποια ζητήματα όσον αφορά την ε, ε, διακυβέρνηση για τα θέματα τη χρηματοδότηση, γιατί κατόρθωσε το Κοινοβούλιο να καταγαγει κάποιε σημαντικέ νίκε. νίκες. Πρώτα-πρώτα έχουμε περισσότερη διαφάνεια σε όλου του ε, τομεί εργασία ε, τη σχετική υπηρεσία. και επίση είμαστε πλήρω μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτή η υπηρεσία προηγουμένω ήταν γνωστή ω το εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς, έτσι ήταν το όνομα. Και τώρα ο τίτλος θα είναι ε, <clears throat> η Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Συνωματικής Διοκτησίας. EU και οπότε ε, προσπαθήσαμε τα σχετικά τέλη να τα μειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο χωρίς να πειράξουν τα εθνικά συστήματα. Επίσης αυξήσαμε τη χρηματοδότηση τη σχετική με την συνεργασία μεταξύ της ε, υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών υπηρεσιών και έτσι έγινε αυτό που λέμε soft harmonization και επίσης έγινε και το capacity building, δηλαδή βοηθήσαμε τις δυνατότητες των ε, εθνικών υπηρεσιών. Και όπως είπαμε επανειλημμένα στο παρελθόν, όλα τα χρόνια, ε, αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι εξυγχρονισμό, όχι επανάσταση. Ε, πρόκειται επομένως για κάτι το οποίο χρειαζόταν και με το παραπάνω όσον αφορά το δίκαιο των σημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι δε ότι αυτό θα μας οδηγήσει εις ε, έναν κοινό σκοπό που έχουμε, δηλαδή το πώς θα έχουμε περισσότερη ανάπτυξη και ευημερία στην Ευρώπη, κάτι το οποίο τη σήμερα ημέρα το χρειαζόμαστε τόσο πολύ. Θεωρώ δε ότι οι συνάδελφοι πρόκειται να ε, επιψηφίσουν αυτό το κείμενο στο οποίο συμφωνήσαμε. Σας ευχαριστώ για την ε, βοήθειά σας και σας ευχαριστώ για τα όσα τόσο επικοδομητικά και ζωηρά συζητήσαμε. Καλή συνέχεια. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος, την κυρία Βίξτρομ. Ε, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους έλαβαν μέρος σε αυτήν τη συζήτηση, αλλά και την ε, κυρία Πίτροπο. Εδώ κλείνει αυτή η κοινή συζήτηση. Θα ψηφίσουμε το κείμενο αυτό αύριο. Το επόμενο θέμα τη διατάξεως είναι η δήλωση της Επιτροπής σε σχέση με την προστασία των θυμάτων της ε, τρομοκρατίας. Θα δώσουμε τώρα τον λόγο στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Μπιενκόφ,